Κοινοβουλίου υπέγραψε από κοινού με τον πρόεδρο του Συμβουλίου τον κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ο τίτλος εν λόγω πράξη θα δημοσιευτεί στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης. Η Επιτροπή Περιβάλλον